Uh, Αγαπητοί φίλοι, θα αρχίσουμε σύντομα να ψηφίζουμε, οπότε καθίστε και ετοιμαστείτε για την ψηφοφορία. Thank you. Uh, Αρχίζουμε λοιπόν. Και ψηφίζουμε μαζί οι Επιτροπές Απασχόλησης και Πολιτισμού Έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Την έκθεση για τις καλύτερες υπηρεσίες όσον αφορά τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα του Europa Super. μάλλον είπα ηλεκτρονική διορθώνει πρόεδρος, οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Εντάξει, αφήνουμε ανοιχτή ακόμα την ψηφοφορία γιατί βλέπουμε ότι έρχεται κόσμος, προσπαθεί να καθίσει, να βρει την κάρτα του για να ψηφίσει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα μπορώ να κλείσω την ψηφοφορία. Καλώς. Ωραία. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. προχωράμε στο επόμενο θέμα που είναι η εκλογή των εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά ίσως η Επιτροπή Πολιτισμού θέλει να πει δύο λόγια για την ψηφοφορία που μόλις κάναμε πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ήταν μια πολύ σημαντική ψηφοφορία, έτσι. Έχετε το λόγο, κύριε Κάμερφαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Μαϊτέ. Πρώτα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την θαυμάσια συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών μας. Το αποτέλεσμα που επιτύχαμε στον τριμερή διάλογο είναι πολύ θετικό. Και ασφαλώς δεν ήταν πάντα εύκολο, δεν ήταν πάντα εύκολη υπόθεση και γι' αυτό ευχαριστώ τους δύο εισηγητές που νομίζω ότι δούλεψαν καλά, και βεβαίω θέλω όλος ιδιαίτερω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες Ένοντι Καμώνα και την Άννα Μαρία Ριβέρα της Γραμματείας που της Γραμματείας Επιτροπής Πολιτισμού που δούλεψαν πολύ σκληρά για το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν ευχαριστώ τα δύο αυτά πρόσωπα εγκάρδια. Και το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικό. Και με μεγάλη ευχαρίστηση θα συνεχίσω με τη συνεργασία με την Επιτροπή σας. Ευχαριστούμε. Εσεί είστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα, κύριε Μάν, κύριε λοιπόν- Α, κύριε θέλετε και εσεί το λόγο. Παρακαλώ. Ο κύριο Μάν. Ευχαριστώ και ιδίω για την συνεργασία. Δεν είναι και συνηθισμένη μια τόσο αγαστή συνεργασία μεταξύ κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θα επιτύχουμε μεγαλύτερη κινητικότητα, απλούστευση των διαδικασιών Θέλουμε να μπορούν να καταγράφονται οι διάφορες δεξιότητε και προσόντα τα οποία αποκτούν τα πρόσωπα. Ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία και ιδίως μπορέσαμε να δεσμεύσουμε Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι ξεκινήσαμε όλα τα θεσμικά όργανα από διαφορετικές θέσεις. Είναι λοιπόν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και ίσως μάλιστα μπορεί να αποτελέσει και υπόδειγμα για τα πράγματα εκείνα τα οποία δεν μπορούν οι χώρες μέλη να κάνουν μόνες τους, ότι μπορούν να γίνουν καλύτερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Ο κύριος Μάλινοφ τώρα. Ευχαριστώ. Πάντα ευχαριστούμε τη γραμματεία μας, αλλά αυτή τη φορά πιστεύω ότι πραγματικά το έργο τους ήταν πολύ πιο σημαντικό από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις, επειδή η υπόθεση ήταν πολύ δύσκολη. Και τους ευχαριστώ πολύ για την υπομονή τους και για την υπομονή τους να δουλέψουν μαζί μου. Ευχαριστώ και τον κύριο Μαν. Με ιδιαίτερη χαρά συνεργάστηκα μαζί του. Τόσα χρόνια καθόμαστε εδώ δίπλα ένας στον άλλον λόγω αλφαβητικής σειράς αλλά έτσι αποδεικνύεται ότι δεν μπορούμε μόνο να καθόμαστε δίπλα, αλλά μπορούμε και να συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Οπότε περιμένουμε την επόμενη αναθεώρηση του Europass που είναι αναπόφευκτη αλλά θα είναι σίγουρα πολύ πιο εύκολη εξαιτία του τόσο καλού έργου που πετύχαμε σε αυτήν εδώ την αναθεώρηση. Παρόλο λοιπόν που είχαμε μια πολύ δύσκολη εκκίνηση νομίζω ότι καταλήξαμε πολύ θετικά κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι μπορούμε να πετύχουμε συνενέσεις και συμφωνίες ακόμα και όταν ξεκινούμε από θέσεις ε, διαμετρικά αντίθετες με το Συμβούλιο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ωραία, περνάμε στις επόμενες ψηφοφορίες τώρα και αποχαιρετούμε εδώ την Επιτροπή Πολιτισμού. Μυστική ψηφοφορία. Τώρα, για τους εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.